για την ε, εφαρμογή της ε, Οδηγίας 2273 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανθρώπων και γυναικών στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και την πρόθεση και τις συνθήκες εργασίας. Έκθεση που είναι υπε, για την οποία είναι υπεύθυνη η κυρία Τερεζαριέρα Μαδουράη που έχει τέσσερα λεπτά για να κάνει την παρουσίασή της. Κύριε Βουλευτά, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η οδηγία στην οποία αναφέρεται η έκθεση τροποποιεί μία η οδηγία του 78 για το ίδιο θέμα που άλλαξε μετά τη συνθήκη του Άμστερνταμ την ομολογία του ΔΕΚ και, τις νέες, και τη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Ε, ενσωματώνει βασικά στοιχεία στο θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών. Το κείμενο της οδηγίας εισάγει τον ορισμό της έμεσης και άμεσης διάκρισης της και της σεξουαλικής και μη σεξουαλικής παρενόχλησης, υιοθετώντας, προτείνοντας τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μέτρα για να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις με βάση το φύλλο και να προστατεύσουν τα, εργασιακά δικαιώματα. Στα πλαίσια της άδεια μητρότητας ή πατρότητας επιπλέον, πέραν της δημιουργίας ε, δομών προς την ισότητα που ζητούμε να δημιουργήσουν τα κράτη-μέλη, περιλαμβάνουν την δέσμευση των κρατών να ξεκινήσουν και να ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο για να προωθήσουν την ισότητα στο εργασιακό πλαίσιο μέσω συλλογικών συμβάσεων και με ρυθμισμένο τρόπο. Επίση, ενισχύεται ο ρόλο των ΜΚΟ στην πρόθεση τη ισότητα, θεσπίζονται συγκεκριμένα μέτρα κυρώσεων για όσου δεν τηρούν τι νομοθετικέ διατάξει και την εφαρμογή μέτρων προστασία για όσου ε, θέλουν να υποστηρίξουν τα θύματα. Η Κομισιόν αν μπορούσε να ετοιμάσει μια έκθεση δεν, που με βάση την οδηγία θα έπρεπε να γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια, η δουλειά μας ήταν απλή. Ωστόσο, για το λόγο αυτό θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να έχουν εμπρόθεσμα ενσωματώσει την οδηγία. Να το έχουν κάνει καλό και να έχουν δώσει τα στοιχεία ενημέρωση στην Κομισιόν. Δεν είναι αυτή η κατάσταση από την οποία ξεκινούμε ωστόσο. Όταν έλεξε η προθεσμία εφαρμογή τη οδηγία, ε, τα κράτη-μέλη δεν είχαν αναφέρει τα μέτρα που έλαβαν για την υλοποίηση. Η Κομισιόν ξεκίνησε διαδικασία παραπομπή. Τον Μάιο του περασμένου έτου υπήρχαν ακόμα ανοιχτέ διαδικασίε, εκκρεμεί διαδικασίε κατά δύο κρατών μελών. Επιπλέον δεδομένου του περίπλοκου χαρακτήρα της οδηγίας αυτής, η Επιτροπή είχε διαπιστώσει προβλήματα στην ενσωμάτωση σε διάφορα κράτη-μέλη. Ήλπιζε να, να, σώσει πολλά από αυτά μέσω, μέσω, να λύσει πολλά από αυτά μέσω του διαλόγου. Για να υπάρξει ωστόσο μια πλήρη έκθεση, χρειαζόμασταν να έχουμε στοιχεία, περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή μα. Γι' αυτό ζητήσαμε πληροφορίε και από τα κράτη-μέλη. Οι πληροφορίες που μας έδωσε η Επιτροπή και, αυτή, και αυτές που λάβαμε από τα κράτη-μέλη μέσω των οργανισμών πρόσφυσης της ισότητας και των εθνικών κοινοβουλίων και με τις συνεισφορές των συναδέλφων από τις διάφορες πολιτικές ομάδες καταθέσαμε να ετοιμάσουμε την έκθεση αυτή που δίνει μια σαφή ιδέα του πώς γίνεται η διαδικασία ενσωμάτωσης ε, της νομοθεσίας σε κάθε κράτος μέλος. Μετά τις εμπειρίες που είχαμε, θέλω να πω ότι η συνεργασία μεταξύ των εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε καθοριστική σημασία για να μπορέσουν να κάνουμε σωστά τη δουλειά που κάναμε. Αν ε, χωρίς τις πληροφορίες αυτές από τα κοινοβούλια και τους οργανισμούς ισότητας δεν θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε την έκθεση αυτή με την ε, ευρύτητα που περιέχει αυτή τη στιγμή. Ούτε το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε χωρίς και την συνεισφορά τη επιτροπή, ιδίως ε, της επιτροπή Γυναικών του γραφείου μου και των υπηρεσιών της κοινοβουλευτική μου ομάδας. Σε όλες τις γυναίκες αυτές θέλω να, ε, όλες τις γυναίκες αυτές θέλω να τις ευχαριστήσω. Ταυτόχρονα να ευχαριστήσω και τις σκιώδεις εισηγήτριες. Εξ αρχής, ο στόχος μας ήταν ε, να υπάρξει μια συνένεση ε, στην συζήτηση για να έχουμε μια καλή εικόνα της κατάστασης στην οποία ε, υπάρχει η εφαρμογή μιας πολύ σημαντικής οδηγίας που δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά εφόδια ώστε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν την νομοθεσία για, το, την, για την ισότητα στον χώρο εργασίας. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα, ακόμα και σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλη διαφορά, 28,4% ε, σε ό,τι αφορά την, τον αριθμό, το, το ποσοστό των ανδρών και γυναικών αντίστοιχα που εργάζονται. Μην ξεχνάτε επίση ότι οι γυναίκες κατά μέσο όρο λαμβάνουν 15% λιγότερα αμοιβέ, λιγότερο μικρότερη αμοιβή από ότι οι άνδρες. Αν δεν αν μπορέσουμε να αυξήσουμε την επίγνωση της ανισότητας αυτής, σίγουρα θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ Τερέζα. Η Επιτροπή. Κυρία Βασιλείου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Η Κομισιόν δέχεται την πρόταση του Κοινοβουλίου για την οδηγία αυτή και ευχαριστούμε την κυρία Μαντουρέλα για τη σκληρή τη εργασία. Η οδηγία 2002 κάθετος 73 τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση τη άνηση μεταχείριση των φύλων, την πρόσβαση, στην εργασία και την επαγγελματική εκπαίδευση και την προώθηση των καλύτερων συνθηκών εργασία. Έχει δε σημαντικά βελτιώσει την κοινοτική νομοθεσία στο θέμα αυτό με σαφέστερε διατυπώσει και ορισμούς του, των διαφόρων τύπων άνησης μεταχείρισης. Συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για τις εγγύους και για τις, εγγύους που παίρνουν γονική, για τις γυναίκες που παίρνουν γονική άδεια για να διασφαλιστεί έτσι η ισότητα των φύλων στον τόπο εργασίας και να καθοριστούν και εργαλεία και σώματα ελέγχου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν μεγάλες ανισότητες ακόμη μεταξύ ανδρών και γυναικών στους τόπους εργασίας. Τονίζει, εφιστά την προσοχή των χωρών μελών στην Επιτροπή στους κοινωνικούς εταίρους και στην κοινωνία των πολιτών προς τις οδηγίες που ισχύουν για το θέμα αυτό και τονίζει ότι πρέπει να εφαρμοστούν απόλυτα, πλήρως. Γι' αυτό μπορεί να συνεισφέρει σε καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και σε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της κοινωνικής νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση ανδρών αλλά και γυναικών. Ως θεματοφύλακας των συνθηκών οικομισιών θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των οδηγιών στα κράτη-μέλη. Η ιδέα συνέχιση του διαλόγου με τα κράτη-μέλη και οι πιθανές προσφυγές τις οποίες θα κάνουμε για να διασφαλιστεί η ισότητα είναι κάτι το οποίο δεν θα διστάσουμε ποτέ να πράξουμε η Κομισιόν θα εγκρίνει δε μια σχετική έκθεση το κατά το πρώτο ήμιση του έτους για την εφαρμογή των οδηγιών σε όλες τις χώρες μέλη και θα υποβάλει τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία μου. Η έκθεση θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Τελειώσαμε συνάδελφοι την σημερινή συνεδρίαση. Αύριο θα έχουμε τη νέα συνεδρίαση, 13 του μηνός, 9 με 1, ως συνήθως, 3 με 7 και 9 με 12 τη νύχτα. Η ημερήσια διάταξη είναι στο σχετικό έγγραφο και